Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Τα χθεσινά συνοπτικά πρακτικά έχουν διανεμηθεί και θα πρέπει να τα εγκρίνουμε. Και σας ερωτώ αν έχει κάποιος ε, παρατηρήσεις, αντίρρηση, κάτι να επισημάνει για τα πρακτικά. Όχι, εγκρίνονται λοιπόν τα χθεσινά συνοπτικά